θέμα το αναγνώρισαν πολύ ότι είναι ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε στο σημείο αυτό και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και η εξωτερική εκπροσώπηση του ευρώ. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Επίτροπο, τον κύριο Ρεν. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Uh, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα που θέσατε. Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Δούνου του στις 20 Μαΐου που αποσαφηνίζει τη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Διευθυντή του. Συμφωνούμε ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ανοιχτή, διαφανής και να βασίζεται σε αξιολογικά κριτήρια. Γιατί υπάρχουν κατάλληλοι ικανοί υποψήφοι από όλε τις χώρες του για να, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη όλα τα προσόντα που διαθέτουν. Οι χώρες της Ένωσης συμφώνησαν να υποστηρίξουν τον αξιότερο, εκείνον που θα πληρεί τα υψηλότερα κριτήρια και προσόντα που απαιτούνται στη θέση αυτή. Ένας τέτοιος υποψήφιος πρέπει να έχει επιδείξει τις ικανότητες του και την θέλησή του να καθώς και τη γνώση του της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κατάστασης. Η Κομισιόν υποστηρίζει τη συμφωνία και επίσης την υποψηφιότητα της Υπουργού κυρίας Χριστίνας Λαγκάρντα που είναι ικανή και έμπειρη υποψήφια που έχει κερδίσει το σεβασμό όλων των εταίρων μας στη διεθνή κοινότητα. Δεν έχει μόνο μεγάλη γνώση της ευρωπαϊκής οικονομίας, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό προσόν στην εποχή μας, αλλά και μεγάλη εμπειρία στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, παραδείγματος χάρη στη διαχείριση που ε, επέδειξε του ΓΑΜΑ 20, του ΖΙΤΑ 20, Πέρυσι είχε συμφωνηθεί στο z 20 στην Κορέα να μειωθεί η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δουνουτού κατά δύο θέσεις για να αυξηθούν οι δυνατότητες εκπροσώπησης των αναδειωμένων οικονομιών αγοράς. Έτσι, Ενώ όλα αυτά σχετίζονται με το γενικότερο θέμα της μεταρρύθμισης της λειτουργίας του Ταμείου, δεν σχετίζεται ακριβώς και απόλυτα με το πρόσωπο του Γενικού του Διευθυντή. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κοινό συμφέρον της Ένωσης και των χωρών μελών της να κινηθούμε προοδευτικά προς μία ενιαία έδρα της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο εκεί, προοδευτικά είπα. Κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, εγώ έχω δεσμευτεί υπέρ της μεταρρύθμισης για μια καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση και εσωτερικά και εξωτερικά. Και θα προτιμούσα να εφαρμοστεί η δοκιμασμένη μέθοδος του Ζαν Μονέ, δηλαδή η πρόοδος να σημειώνεται στη βήμα το βήμα, με περισσότερα και μικρότερα βήματα δηλαδή. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να καταλήξει η μεταρρύθμιση της εσωτερικής μας διακυβέρνησης που είναι απόλυτα απαραίτητη και επίγουσα και αυτό θα αποτελέσει πολύ σημαντική πρόοδο για το δεύτερο βήμα της εξωτερικής μας εκπροσώπησης που θα είναι και αυτό σημαντικό βήμα για την ε, βελτίωση της διεθνούς διακυβέρνησης. Ένα μεγάλο βήμα τη φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Όταν ο Γενικός ε, Διευθυντής του Διευθυντικού Ταμείου είχε υποβάλει την υποψηφιότητά του, ο προηγούμενος ε, του είχαμε υποβάλει πολλά ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του Διευθυντικού Ταμείου. Εν τω μεταξύ διαπιστώσαμε και ποιες μπορεί να είναι οι διεθνείς ε, αλληλεπιδράσεις και μάλιστα σε περιβάλλον διεθνούς κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας πλέον και κατανοούμε πλέον όλοι πόσο σημαντικό είναι να είναι είναι πολύ, πολύ ε, ικανή η πραγματογνωμοσύνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γιατί μπορεί να βοηθήσει πραγματικά και θέλουμε στα επόμενα χρόνια να ε, είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει τη δυνατότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παίξει ε, σημαντικό ρόλο στην διεθνή σκηνή και σε αυτήν την κρίση του ευρώ δυστυχώς Δυστυχώς ε, έχουμε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και πολλά λυπηρά γεγονότα έχουν λάβει χώρα. Ε, λέω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει ο νέος Γενικός Διευθυντής να ξέρει καλά και την κατάσταση στην Ευρώπη. Λέτε ότι θα πρέπει να βασιστούμε στην αξία του υποψηφίου, αλλά να μην ξεχνούμε ότι είναι εξαιρετική η υποψήφια που έχουμε εμείς και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελπίζω μάλλον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα ε, θα στηρίξει αυτήν την υποψήφια. Πάντως, κυρίως σε περιβάλλον και σε χρόνο κρίσης είναι σημαντικό να έχουμε ε, ένα άτομο με, ιδιαίτερες, ε, με ιδιαίτερη ποιότητα και ιδιαίτερες ικανότητες ε, και μάλιστα γυναίκα ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Λαγκάρτ ξέρουμε ότι έχει σημαντική εμπειρία και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού. Πρόκειται για μια εξαιρετική υποψήφια και ελπίζω ότι με τη στήριξή μας και με τη δική σας στήριξη θα μπορέσουμε να ε, δούμε την κυρία Λαγκάρντε στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Η κυρία Μπερές για τέσσερα λεπτά εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αναρωτιέμαι πραγματικά γιατί θέλησατε να κάνετε αυτή τη δήλωση. Ακούω την παρέμβασή σας. Ακούσα. Σας άκουσα να λέτε ότι σε τελική ανάλυση εμείς έχουμε όλοι ξεκινήσει στην αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης και την εκπροσώπηση και το θέμα της εκπροσώπησης ζώνης του ευρώ θα την αντιμετωπίσουμε αργότερα. Επιτρέψτε με να μην συμμερίζομαι την προσέγγισή σας, γιατί νομίζω ότι μία από τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το θέμα της εξωτερικής της εκπροσώπησης για τη ζώνη του ευρώ βλέπουμε ότι ο πόλεμος των νομισμάτων μπορεί να σαρώσει όλες τις προσπάθειες που ζητούμε από τους λαούς στη ζώνη του ευρώ μέσα στα πλαίσια της λιτότητος και της επαναφοράς της ομαλότητος για το δημόσιο χρέος. Η Ευρώπη λοιπόν δεν μπορεί να είναι τόσο απαιτητική στο εσωτερικό της και να μην δίνει σημασία για τη θέση του νομίσματός της στο εξωτερικό το οποίο κινείται από εδώ και από εκεί στο έλεος των αγορών. Αν δεν υπάρξει λοιπόν εξωτερική εκπροσώπηση δεν μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο εκεί. Γι' αυτό διαφωνώ μαζί σας. Ξέρω ότι είναι δύσκολος ο ρόλος αυτός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια έχει υποστηρίξει την ιδέα ότι πρέπει να κινηθούμε προς μια ενιαία εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το, στις, τη ζώνη του ευρώ μάλλον και ιδιαίτερα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν ο Ντόμινικ Στροσκάν ανέλαβε τα ύπατα αξιώματα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν πολύ διαφορετικά τα, τα θέματα. Υπήρχε και το θέμα αυτό της εναλλαγής στην εξουσία, στην κορυφή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είχαμε τονίσει τη σημασία να υπάρχει ένας Ευρωπαίος εκεί, αλλά έχουν αλλάξει πια τα πράγματα. Η... Το μέρος που είναι αποφασιστική η δράση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι σήμερα η Ευρώπη. Και τίθεται και το θέμα τις δράσεις των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών στις ΗΠΑ που δεν είναι πια ουδέτερη η δράση τους σε σχέση με την κρίση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να τεθεί λοιπόν το θέμα αυτό και αυτό είναι ένα θέμα θα πρέπει να συζητηθεί και μέσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά μας δημιουργούν ένα τοπίο που είναι πολύ πιο πολύπλοκο από το απλό θέμα του αν θα πρέπει να είναι το α ή το β άτομο το οποίο θα πρέπει να προεδρεύει του διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Εμείς ως Ευρωπαίοι φυσικά θα πρέπει να έχουμε μια εκπροσώπηση. Να παίζουμε ένα σημαντικό ρόλο σε ένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς φορείς. Αλλά το πραγματικό ερώτημα για μένα είναι τι είδου πολιτική θέλουμε να ακολουθήσουμε στο διεθνές στερέωμα. Τι εντολή θα πρέπει να έχει ένα Ευρωπαίο που μας εκπροσωπεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. λαμβάνοντα υπόψη την τι ενέργειε που γίνονται στο εσωτερικό μα, λαμβάνοντα υπόψη την επίπτωση των αγορών στην εσωτερική κατάσταση τη Ευρώπη σε ό,τι αφορά τι επενδύσει, την κερδοσκοπία, τι θέσει απασχόληση. Πιστεύουμε περαιτέρω ότι ανεξάρτητα από το άτομο το οποίο θα διευθύνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο καθήκον. Το να μην καταστρέψει όλη την πρόεδρο, όλη την πρόοδο που επετέφθη από τον Ντομινίκ Στροσκάν, ο οποίος κίνησε προς τα εμπρός την ε, συνένεση στη Ουάσιγκτον. Βλέπουμε τώρα να, να σκληραίνει η αντιμετώπιση και να υπάρχουν οι παραχωρήσεις. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Τέλος, το να μπορέσει να ενσωματωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβει υπόψη και η Ευρώπη αν έχουν κάποιο υποψήφιο θα πρέπει αυτός ο υποψήφιος να μπορέσει να υποστηρίξει μια καλύτερη παγκόσμια διακυβέρνηση για τα οικονομικά θέματα που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε και την οικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο για την ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων, ο κύριος Σμιτ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε ότι ο κύριος Τροσκάν αυτή τη στιγμή είναι υπόδικος για, μια, για ένα σοβαρό αδίκημα. Και αυτό έχει ρίξει τη σκιά του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μέσα στις συνθήκες αυτές είναι σημαντική η επιλογή του ατόμου που θα διαδεχθεί τον κύριο Στροσκάν για το κύρος και του οργάνου αυτού. Εμείς θεωρούμε ότι η κυρία Λαγκάρτ είναι ένα ιδιαίτερα ικανό άτομο και υποστηρίζουμε πλήρως την υποψηφιότητά τους και ελπίζουμε θα έχει την πλήρη υποστήριξη και της Κομισιόν και των κρατών μελών. Γιατί όμως δεν μπορούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία για τον διορισμό αυτού του εκπροσώπου. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ την Ευρώπη να έχει μεγαλύτερο κύρος. Αν είχαμε μια τέτοια διαδικασία, μια κοινή διαδικασία και αν η Κομισιόν είχε τη δυνατότητα να παίζει ρόλο σε αυτή τη ε, διαδικασία επιλογής, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μεγαλύτερη ακτινοβολία προς τα έξω. Το λέει και η συνθήκη της Λισαβόνας, ότι το άρθρο 238 τονίζει τη σημασία μιας κοινή εκπροσώπησης προς τα έξω. Γιατί εμείς δεν ακολουθούμε όμως αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν ενισχύουμε περισσότερο την εξωτερική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε και η κυρία Μπέρες, Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη σαφήνεια σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια ενιαία εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα είναι και στεναρή. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο να παίζει το ρόλο του <clears throat> επενδυτή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αντιμετώπιση τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι πραγματικά παγκόσμια, δεν είναι οικουμενική και αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Σουέμπερν έχει το λόγο τώρα για δύο λεπτά από τις Ευρωπαίους Συντηρητικούς Μεταρρυθμιστές. In today's uncertain economic σε αυτό το αβέβαιο ε, οικονομικό κλίμα και πλαίσιο είναι βέβαιο ότι θα πρέπει και μέσω του Διεθνούς Ομιλωτικού Ταμείου να βοηθηθεί η διεθνή σταθερότηση. Ε, δεν υπάρχουν χώρες ε, οι οποίες ε, αρέσκονται στο να κάνουν συμβολικές δηλώσεις. Όμως το ΔΝΤ δεν είναι σύμβολο. Αβοηθάει στη διαχείριση της οικονομίας και έχει την ικανότητα να μεταφέρει αυστηρές προϋποθέσεις προς τις οικονομίες. Το υπέρ, το σύνε της κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ δεν είναι ότι είναι Ευρωπαία, είναι ότι έχει έχει την δυνατότητα να ηγηθεί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχει την ε, ικανότητα να διαχειριστεί ε, ε, τα δέσμες μέτρων που θα επιτρέψουν σε χώρες οι οποίες βρίσκονται σε δινή οικονομική κατάσταση να ξεπεράσουν τις συμπληγάδες και επομένως να τις βοηθήσει να βρουν μια ευτυχή λύση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, ότι δεν υπάρχει μόνο η σημερινή δινή οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι τα μελλοντικά προβλήματα τα οποία ενδεχομένω θα αντιμετωπίσει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και επομένω θα πρέπει ε, να, είμαστε βέβαιοι ότι μέσω και του νέου Γενικού Διευθυντού ε, θα συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και στο μέλλον. Όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση του ευρώ, αυτή δεν πρέπει να γνωρίζει εθνικά σύνορα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντονιστούν οι εθνικές πολιτικές ε, και ε, να ε, υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διασύνδεση των πολιτικών έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα νομοθετικά κενά και σίγουρα τα κενά αυτά να μην δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση του ευρώ. Ε, υπάρχουν ε, σημαντικές διαφορές ε, μεταξύ των χωρών της ζώνης ευρώ και βεβαίως ακόμα μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών της ζώνης ευρώ και των μη. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σε προσεκτικοί να μην υπάρχουν άλλες απόψεις. Ομάδα των Πρασίνων, ο κύριος Λάμπερτς για δύο λεπτά παρακαλώ. Δυόμιση λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτον, ε, να μιλήσω για τη διαδικασία, όπως και στην άνθρωπο ε, Σμιτ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, η θέση του Γενικού Διευθυντή του ΔΕΛΤΑΝΗ ΤΑΦ. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές, ακόμα και βλέποντας πόσο δύσκολα επιλέγεται ένας απλός διευθυντής σε μια εταιρεία, πραγματικά μας αφήνει λίγο έκπληκτους ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή του νιτάφ και δεν είναι δυνατόν σε, δια, σε καθεστώς αδιαφάνειας να συνεδριάζουν κάποιοι επικεφαλής κυβερνήσεων και να λένε ε, μάλλον να προωθήσουμε αυτόν ή τον άλλον στη θέση του Γενικού Διευθυντή ε, και επομένως ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, και ε, σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς δεν είχαμε τη διαφάνεια και τη συζήτηση που είχαμε. Βεβαίως δεν είστε εσείς υπεύθυνο, αλλά παρόλα αυτά στο μέλλον θα πρέπει να το ξέρουμε. Ε, δεύτερον, και εδώ θέλω να απαντήσω στην κυρία Σουίνμπεργκ, ε, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να απαντήσουμε και σε εσά κυρία Σουίνμπεργκ και στον κύριο Φάραζ, σε ανθρώπους δηλαδή που θεωρούν εσφαλμένα ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει επίπτωση ας πούμε στις διεθνείς αποφάσεις. Είπε η κυρία Σουίνμπερν ότι θα πρέπει εναρμονισμένα και με μία φωνή ε, να μιλεί η Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν να ακούσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την θεϊκή χοροδία των αρμονικών φωνών. Γιατί ο καθένας εκπροσωπεί τους, του, τους δικούς του εκλογείς. Ε, γιατί υπάρχουν μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, ε, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλες μικρότερες χώρες και επομένως νομίζω ότι βαυκαλίζεστε εάν νομίζετε ότι όλε αυτέ οι χώρε μπορούν να μιλούν με μία φωνή. Ε, τρίτον, η θέση Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντιμετώπιση της κρίσης. Επιστρέφω σε εσά, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι σε όλε τι συζητήσει που γίνονται στι διάφορε τρόικα που επισκέπτονται τι χώρε, τελικά, τελικά είναι το διεθνέ Νομισματικό ε, Ταμείο ε, είναι αυτό το οποίο δίνει τι πιο λογικέ λύσει. Και λυπούμε που το λέω γιατί είχε δαιμονοποιηθεί το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο δεκαετία του 80 και του 90 και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πάντως δεν μπορούμε σαν Ευρωπαίοι να συνεχίσουμε αυτή την ε, ε, κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμπερτ. Ο κύριος Κλούτε έχει το λόγο για 1,5 λεπτό από την ε, ε, Ευρωπαϊκή Αριστερά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν πρόκειται για άτομα. Πρόκειται για μια διαδικασία επιλογής. Εγώ εντυπωσιάζομαι που υπάρχει μονάχα μια απάντηση σε αυτή τη διαδικασία ότι η Αμερική και η Ευρώπη πρέπει να διαμοιράζουν τις θέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή οι ισχυρότεροι όμιλοι στον κόσμο μοιράζουν την πίτα μεταξύ τους τον έλεγχο της ε, παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό, δεν είναι φεδεραλισμός. Κατά τη δική μας άποψη, η αποχώρηση του Ντομινίκ Στροσκάν είναι και μια ευκαιρία ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια εκβάθρον τροποποίηση της διαδικασίας για το διορισμό των υπευθύνων στο επίπεδο αυτό, ώστε να γίνεται με έναν τρόπο ο θα έχει να κάνει με διαφάνεια και με πραγματικά προσόντα και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν ζητήσει πάρα πολλές, μικρο, πάρα μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και να εξασφαλιστεί και μια πλειοψηφία η οποία δεν είναι μονάχα η πλειοψηφία των μετόχων του Διεθνούς Ταμείου, αλλά μια ευρύτερη πλειοψηφία. Μια τέτοια αλλαγή της διαδικασίας σημαίνει και μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί έχουν αλλάξει πια οι διεθνείς ισορροπίες, υπάρχουν και πολλές αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν την εμπειρία τους στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και επομένως το δούνου του θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει και κίνηση προς τη μείωση της ένδυας και της διεθνούς ανισότητας. Κύριος έχει το λόγο τώρα για δύο λεπτά. Κύριε Ρεν, δεν βλέπω το χάρτη του, τη χάρτα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λέει να μειωθούν οι ανισότητες, να αυξηθεί η ανάπτυξη, να βοηθήσει οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε προβλήματα μπαίνουν στι χώρε και οδηγούν σε μια ανταγωνιστική υποτίμηση. Δεν λέει πουθενά ότι ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πέρα για να υποστηρίξει πολιτικά πειράματα. Αυτό έκανε και ο Ντόμινικ Στροσκάν. Χρησιμοποίησε το δούνου του για να βοηθήσει να διασώσει το κλειδονιζόμενο και καταστρεφόμενο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και τώρα θέλετε να το επαναλάβετε αυτό με το να βάλετε την Κριστή Λαγκάρτ να συνεχίσει αυτά τα οποία θα κάνει ο Ντομινίκ Στροσκάν. Ένα άλλο μέλος της ευρωπαϊκής ελίτ, ένα ευρωπαϊκό, ένα κάποιον ο οποίος υποστηρίζει αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο, επειδή έχει τέτοιε τάσεις, είναι ο χειρότερος υποψήφιος. Δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγάγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να είναι μονάχα οι φορολογούμενοι τη ε, ζώνη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο ο κόσμο στην πραγματικότητα που να υποστηρίζει τη ζώνη του ευρώ τη στιγμή που το ελληνικό πρόβλημα γίνεται χειρότερο κάθε μέρα. Βλέπουμε ότι όχι μονάχα θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα, ότι όχι μονάχα προχωρούμε για μια τέταρτη διαδικασία διάσωσης, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τεθεί σε αμφιβολία με όλα αυτά που έχουν γίνει. Δεν μπορείτε λοιπόν να συνεχίζεται να σωρεύεται χρέη επί χρεών. Έχουμε φτάσει στο σημείο που μετά από μερικές εβδομάδες μπορεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι αφαιρέγγια. Ίσως η κυρία Λαγκάτ μπορεί να βοηθήσει να την διασώσετε. Νομίζω ότι είναι λοιπόν μια λανθασμένη επιλογή. Η διεθνή κοινότητα κάποια στιγμή σας, θα σας πει φτάνει. Όχι ακόμα. Δεν το έχει πει αλλά θα το πει. Τώρα ερχόμαστε στους άλλους εγγεγραμμένους ομιλητές. Τον λόγο παίρνει ο κύριος Γκουζές για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ θα εκπροσωπήσω και την κυρία Λούριν και τον κύριο Βερέγκ που δεν είχαν άλλο χρόνο ομιλία, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω το σύνολο του αθροίσματο του χρόνου ομιλία. Θέλω να υπενθυμίσω, όπω έκαναν και άλλοι, ποια είναι η διαδικασία επιλογή που έχει ήδη αρχίσει. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφράσει μια ενιαία θέση και στεναρή που να συμφωνεί με, με την οποία να υπάρξει, από την οποία να υπάρξει συμφωνία και από τα κράτη-μέλη και από την Επιτροπή. Με την εξαίρεση του κ. Φαράτζ όλοι συμφώνησαν ότι η ισορροπία που υπήρχε μέχρι τώρα μεταξύ Ένωσης και ΕΠΑ πρέπει να συνεχιστεί και από τον καινούργιο Γενικό Διευθυντή καθώς και σε συνεργασία με τη Διεθνή Τράπεζα. Κατανοούμε ότι οι αναδυόμενες χώρες, οι δύο σημαντικότερες από αυτές, θέλουν να παίζουν περισσότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και είναι επίση σημαντικό να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση της διευθέτηση, της οικονομικής διαχείρισης όπως υπενθύμησε και ο κύριος επίτροπο. Αλλά είναι ίσως πολύ νωρί για να ζητήσουμε ήδη ριζικές μεταβολές σε βάθος. Ένας ευρωπαϊκός υποψήφιος μόνον έχει αναλάβει πραγματική καμπάνια συνεννόησης με τα κράτη-μέλη, μία υποψήφια μάλλον, που έχει τα απαραίτητα προσόντα, την πολιτική εμπειρία, την ηθική αξιοπιστία, τον έλεγχο της αγγλικής γλώσσης και όλα αυτά την καθιστούν κατάλληλη υποψήφια για Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Ταμείου διαθέτει συνένεση και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο το όργανο αυτό. Πρέπει με την ε, εθελοντική της ε, αποφασιστικότητα να κάνει ό,τι μπορεί και να τη στηρίξει η Ένωση. Την κυρία Χριστίνα Λαγκάρντα. Ο επόμενος συγγεγραμμένος ομιλητής είναι ο κύριος Σικλούνα, αλλά επειδή απουσιάζει θα αντικατασταθεί από την κυρία Μπερές, επειδή είναι από την ίδια πολιτική ομάδα. Δύο λεπτά κυρία Μπερές έχετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βρίσκω ότι υπάρχει ένα παράδοξο στη συζήτηση αυτή. Στην ουσία, ανάμεσα στο, στη Διεθνή Τράπεζα και το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, κυρίως λέμε να μην αλλάξει τίποτα. Ε, εμείς οι Ευρωπαίοι θέλουμε και πρέπει να θέλουμε να λειτουργήσει ε, αυτή η πολυμερή ε, σχέση εάν δεν λειτουργήσει η σχέση αυτή με τους εκπροσώπους των, του G20 να συμμετέχουν σε διάφορες θέσεις. Θα πρέπει να δούμε την δυναμική εξέλιξη της ε, κατάστασης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαφνικά κινητοποιηθήκαμε όλοι για να οριστεί μια Ευρωπαία ε, στην ε, κορυφή του Δέλτα αλλά δεν έχουμε την ίδια, τον ίδιο ίστρο για να πούμε ότι πρόκειται για ένα ακόμα βήμα για την εξωτερική εκπροσώπηση του ευρώ. Γιατί ε, θέλετε οπωσδήποτε να ορίσετε Ευρωπαία επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εάν δεν αυτό δεν αποτελεί αυτό ένα ακόμα βήμα για την εξωτερική εκπροσώπηση του ευρώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί, θα πρέπει να ξέρουμε τι λέμε και να είμαστε βέβαιοι ότι το σύστημα αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει και στο μέλλον. Όσον αφορά την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση, το Διεθνέ Ομισματικό Ταμείο έχει μείζωνα ρόλο, όχι μονάχα ε, σε σχέση με το ε, ευρωπαϊκό χρέο και όσον αφορά ευρωπαϊκέ χώρε, οι οποίε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρέου, αλλά ε, πέρα από τη σταθερότητα της αγοράς ε, το ΔΝΤ ε, πρέπει να συμβάλλει στην διόρθωση των παγκοσμίων ανισορροπιών και επομένως ε, αυτό είναι ένα θέμα παγκόσμια διακυβέρνηση, το οποίο φαίνεται να μην βάζεται καθόλου στη ζυγαριά. Και εμείς σαν σοσιαλιστές λέμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι χρήσιμο για να παίξει ρόλο στην παγκόσμια διακυβέρνηση έτσι ώστε να βοηθήσει στην εξάλληψη των ανισοτήτων. Ευχαριστώ. Κύριος Λε Ιαρίκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Merci, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ δεν θα παραγνωρίσω, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να επιλεγεί ο επόμενος διευθυντής του Διεθνής Νομισματικού Ταμείου. Το πιο σημαντικό όμως για τους λαούς είναι ποιο ρόλο θέλει να παίξει αυτός ο διεθνής φορέας στο μέλλον για να μπορέσει να μας βοηθήσει να βγούμε από τη μεγάλη νομισματική και δημοσιονομική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Χρειάζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δημοκρατικοποιηθεί και να υποστηρίξει την ανθρώπινη ανάπτυξη, την απασχόληση, την εκπαίδευση. Θα πρέπει να σταματήσει η δυνατότητα των ΗΠΑ να έχουν βέτο. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των αναπτυσσομένων και αναδιωμένων χώρων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την κερδοσκοπία και να αποτελέσει ένα σημαντικό ε, πυλώνα σταθερότητος για τις ε, αγροτικές αγορές και να αντιμετωπίσει τους φορολογικούς παραδείσους και τις κερδοσκοπίες, να μπορέσει λοιπόν να δημιουργήσει ένα νέο εγχείρημα ενός παγκοσμίου νομίσματος για την ισορροπία και τη συνεργασία και όχι ανταγωνισμούς και συγκρούσεις περιοχών νομίσματος. Πρέπει λοιπόν οι λαοί να ζουν καλύτερα και όχι να τους εκμεταλλεύονται οι τραπεζίτες. Ο επόμενος εγγεγραμμένος ομιλητής, ο κύριος Λάγκεν, δεν είναι στην αίθουσα και θα πάρει το λόγο αμέσως η κυρία Τούν Ουντ Χόχενστάιν για δύο λεπτά παρακαλώ. E, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς Μιλάμε εδώ για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόνο στα πλαίσια της υπόθεσης που γνωρίζετε όλοι, της υπόθεσης Δομινίκ Στραουσκάν. Εδώ είναι όμως θέμα του κύρους του οργανισμού αυτού, αλλά και κύρους ενός Ευρωπαίου πολιτικού που είχε καταλάβει αυτή την τόσο σημαντική θέση. Ελπίζω να πάψουν κάποτε οι συμπεριφορές που γνωρίζετε όλοι και είναι το μόνο θετικό στοιχείο της υπόθεσης αυτής. Πρέπει να αγωνιστούμε για το κύρος και την εικόνα του Δουνουτού. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υποβάλουμε υποψήφιο με πραγματικές ικανότητες. Κάποιον δηλαδή που να είναι σε θέση να επιφέρει ηρεμία και στις αγορές και στο όργανο γιατί αλλιώς θα βλαφτεί ακόμα περαιτέρω η αξιοπιστία του. Η κυρία Χριστίνα Λαγκάρντ θεωρήθηκε ως η καλύτερη υπουργό Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2009. Διαχειρίστηκε πολύ καλά το Z20 όπως είπε και ο Επίτροπος. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία ότι έχει προσόντα και μπορεί να παίξει το ρόλο του γενικού, της γενικής διευθυντρίας του, του, ιδίως στα πλαίσια αυτής της, της τωρινής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επομένως δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή να τοποθετήσουμε Ευρωπαίος στη θέση αυτή και μάλιστα άνθρωπο που να κατανοεί τις ε, πραγματικότητες της κρίσης και ξέρουμε ότι η κυρία Χριστίνα Λαγκάρτε με τα προσόντα και την εμπειρία της διαθέτει τη γνώση αυτή. Έχει ήδη διαχειριστεί σημαντικά διεθνή θέματα επαναλαμβάνω για τέταρτη φορά έχει μεγάλη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρόκειται να ξεχάσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Το είπε και η ίδια, εάν επιλεγώ θα αφιερώσω όλη μου την εμπειρία, το χρόνο και τις ικανότητές μου ως νομομαθούς και οικονομολόγου καθώς και γυναίκας στην υπόθεση αυτή της αξιοπιστίας του οργάνου. Ευχαριστούμε. Έχουν ζητήσει το λόγο δύο συνάδελφοι. Πρώτος ο κύριος Φερέρα. Παρακαλώ για ένα λεπτό κύριε συνάδελφο. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία της αντικατάστασης του Γενικού Διευθυντή του ΔΝΤ δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος που οξύνεται η κρίση του. Αυτή η τροποποίηση σε ένα από τα βασικά στοιχεία του καπιταλιστικού συστήματος δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις εσωτερικές διαμάχες και αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος και επίσης από το θέμα της μετάθμισης του νομισματικού συστήματος και της αντιμετώπισης του παγκόσμιου πολέμου μεταξύ δολαρίου, γεν, ευρώ κτλ. Βλέπουμε όλο και περισσότερο τις συνέπειες αυτού του πολέμου που τις επομίζονται οι φτωχοί και οι εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να παραγνωρίσουμε και την ευθύνη που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι έχουν συμβιβαστεί με τον νεοφιλελευθερισμό, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να μας οδηγήσει να αντιμετωπίσουμε και τις ε, αναδιαθρώσεις των χρεών στην χώρα του ευρώ και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο εναντίον των θεσμικών παρεμβάσεων που έχουν καθαρά απικιακό και νεοπικιακό χαρακτήρα και που οδηγούν σε υψηλότερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ε, η κυρία Τζαβέλα, για ένα λεπτό παρακαλώ κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, από ό,τι φαίνεται ο 21ος αιώνας θα χαρακτηριστεί από τον πόλεμο μεταξύ πολιτικής εξουσίας και εξουσίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Υπάρχουν χώρες στον πλανήτη οι οποίες κυριολεκτικά κυβερνώνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα ανώνυμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι πολίτες των χωρών αυτών άγονται και φέρονται και καθορίζεται η μοίρα τους από τι θα κάνουν οι αγορές. στο πρόσωπο της κυρίας Λαγκάρτ πιστεύω ότι βρίσκουμε μια άξια και ικανή εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής ένωσης με μεγάλο προσόν την εμπειρία που απέκτησε μέσα από όλη αυτή την θυελώδη περίοδο της οικονομικής κρίσης και πιστεύω ότι είναι μια άξια εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. ευχαριστώ. πολύ κυρία τζαβέλα. ο κύριος Ρούμπικ επίσης για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία τεχνική έτσι έχω να κάνω να φτιάξει κάποιο το μικρόφωνο μου που δεν λειτουργεί. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως είναι το σημαντικό είναι η κυρία Λαγκάρτ να πάρει αυτή την ηγετική θέση. Έχει δείξει σαν Υπουργό Οικονομικών της ε, Γαλλίας ότι γνωρίζει τα πράγματα και μπορεί να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να καταφέρουν να δώσουν αυτό το οποίο χρειάζεται η οικονομία μας και γι' αυτό είναι σημαντικό στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων και η αναδιανομή είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό μια μεταρρύθμιση του, της Παγκόσμιας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι μια μεγάλη προτεραιότητα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρε οι οποίες αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικά προβλήματα να έχουν την χρηματοδότηση αλλά και την τεχνογνωσιακή υποστήριξη για να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκουρέδο επίση θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια συζήτηση η οποία παρακάμπτει τα βασικά ερωτήματα, δηλαδή παρακάμπτει το πρόβλημα το πάρα πολύ σοβαρό του καπιταλισμού σε διεθνές επίπεδο και το πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα των χρηματοοικονομικών αγορών που ποδηγετούν και ελέγχουν τις οικονομίες μας και προσπαθούν να επιβάλλουν τους κανόνες τους στις κυρίαρχες χώρες του κόσμου, ανισχύουν και οξύνουν τις διακρίσεις, τις ανισότητες, την καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την καταστροφή των δημοσίων υπηρεσιών, οδηγούν σε μια όξυνση της κοινωνικής, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδυας, όχι μονάχα σε διεθνές επίπεδο για τις, μικρότερες, για τις φτωχότερες χώρες, αλλά ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλά από τα κράτη-μέλη μας. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μια στεναρή θέση για να τροποποιήσει αυτή την κατάσταση, για να σταματήσουν οι φορολογικοί παράδεισοι, να υπάρξει έλεγχο των χρηματαγορών, να υπάρξει επιτέλους τέρμα στην εκμετάλλευση και την αύξηση των ανισοτήτων. θα είναι εδώ η παρεμβάση των συναδέλφων. Ο Επίτροπος θα πάρει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Mr. Commissioner. You have the floor, Mr. Commissioner. Fine, Madam President, uh, honorable members. Uh, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ουσιοδέστατη αυτή συζήτηση. Ε? και διαβλέπω μεγάλη συνένεση στο σώμα για την διαδικασία επιλογής ε, του νέου Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και συμφωνούμε όλοι ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι ανοιχτή, διαφανής και να βασίζεται στην αξιοκρατία. Βλέπω ότι υπάρχει ευρεία, όχι πλήρης, αλλά πάντως ευρεία στήριξη της υποψηφιότητα της κυρίας ε, ε, Λαγκάρντ, την οποία έχουν ήδη ενστερνιστεί ω υποψηφιότητα, λέγω, ε, και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υποψήφια για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Τάφα. Ακούστηκαν διάφορε απόψει στη διάρκεια της ε, συζήτησης. Βεβαίω το Δελτανιτάφα έπαιξε σημαντικό ρόλο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έτσι ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα της κρίσης χρέους ε, σε διάφορες χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πρώην κενικό Διευθυντή Δομινίκης Ροσκάν κατέβαλε μεγάλε προσπάθειε προ αυτή την προσπάθεια. Εξακολουθούν να υπάρχουν βεβαίω κάποιε αναταράξεις όσον αφορά ε, την κρίση χρέους ε, κάποιων ε, χωρών και όσον αφορά την θέση τους στις αγορές, αλλά παρόλα αυτά εμείς έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να ανακάμψει οικονομικά η Ευρώπη. Βεβαίως η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί και επομένως θα αναμένεται και τις επόμενες εβδομάδες περί τα τέλη Ιουνίου να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο Τη της τη της Ευρώπη είναι βέβαιο ότι δεν θα δείτε διαδικασία τύπου πτώχευσης Lehman Brothers στην ε, Ευρώπη. Δεύτερον, είχαμε καλή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, πράγμα όχι απολύτως αυτονόητο όταν αυτή η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο περίπου στα πλαίσια αυτής της μεγάλης χρηματοοικονομικής ε, ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Βεβαίως το κάθε όργανο έχει τη δικιά του φιλοσοφία, έχει του δικιούς του ε, κανόνες αλλά και την ε, δικιά του ανεξαρτησία και επομένως δεν ήταν απολύτω αυτονόητο ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μεταξύ μα αγαστά. Αλλά επεδείχθη ε, πραγματισμός, ορθολογισμός και καλό πνεύμα στην εργασία έτσι ώστε να συγκρατηθεί η κρίση χρέους και να βοηθηθεί η οικονομική ανάκαμψη των χωρών. Συμφωνώ βεβαίως ότι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την εξωτερική εκπροσώπησή μας. Όπως είπε και στις αρχικές μου παρατηρήσεις, είναι τεράστια ε, η ευθύνη ε, που έχουμε και όσον αφορά την μεταρρύθμιση της εσωτερικής οικονομικής ε, διακυβέρνησης και στη διάρκεια του Ιουνίου και πάντως πριν τις καλοκαιρινές διακοπές θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις κατά την έννοια αυτή. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να προσπαθήσουμε, θα πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η απαραίτητη μεταρρύθμιση της εσωτερικής οικονομικής διακυβέρνησης. Μακροπρόθεσμα ο στόχος μας τουλάχιστον για την ε, περιοχή του ευρώ ε, είναι να βελτιώσουμε τη γενικότερη κατάσταση αλλά αυτό σημαίνει ότι ε, βράχει πρόθεσμα ε, θα πρέπει να ε, βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση και στα πλαίσια της Ευρώπης και στους G20 και με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει, λοιπόν έτσι ώστε τα ε, κράτη-μέλη να έχουν καλή ε, αντιπροσώπηση ε, και όσοι εκπροσωπούν την Ευρώπη στους G7, στους G20 και στο Διεθνές Πνευματικό Ταμείο να έχουν κοινού ευρωπαϊκού στόχου. Ναι, βεβαίω έχουν υπάρξει πολλές βελτιώσεις. Ναι, έχουμε πολλά σχέδια για το μέλλον και βεβαίω οπωσδήποτε θα πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά τα τα ε, ζητήματα και θα ξανασυζητήσουμε το θέμα της εξωτερικής εκπροσώπησης του ευρώ. Ε, ο ρόλος των ε, αναδειωμένων οικονομιών είναι σημαντικός και σε σχέση με την ίδια την Ευρώπη και τους πολίτες της Ευρώπης. Αλλά σίγουρα ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε πολύ, καλύτερη, πολύ καλύτερο μέτωπο απέναντι και στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Έληξε η συζήτηση εδώ ε, και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο που είναι εντελώς διαφορετικού περιεχομένου. Είναι η έκθεση του κυρίου Οντί ε, αναφορικά με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης